afternoon, colleagues. Καλησπέρα, συνάδελφοι. The sitting is now resumed. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Παίρνουμε στις ψηφοφορίες. Πολύ άριθμες. Και σας παρακαλώ να συνεργαστείτε για την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους. Έκθεση Εμένοβιτς. Μία ψηφοφορία μία ε, τροπολογία, συγγνώμη, την ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. Απερίφθη. Εγκρίνεται λοιπόν οριστικά η πράξη με βάση τη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Περνώ στην έκθεση Ταραμπελά. Τροπολογία μόνο ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά αρχής προφορία ψήφισαν οι πάντες πέρας και εγκρίνεται. Έκθεση Φλέκενστάιν. Τροπολογία 148 ονομαστικά παρακαλώ άρχεται. Πέρας. Και απερίφθη. Τώρα έχουμε μια σειρά τροπολογιών ε, από αριθμούς έως 135 τσέχτες. στον κατάλογο υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Θα επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για την επαλήθευση πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται όντως. 41 ονομαστικά. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη. 139 ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία της Επιτροπής Φαρθμού 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140D δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 141D δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 150 ονομαστικά. Ε, πέρασε τις προφορίες και απερίφθη. 137 ονομαστικά. Πέρα της ψηφοφορίας Και απερίφθη. 142 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη. 48 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 154 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη 151 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη 152 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη. 143-147 ονομαστικά. Πέρας. Απερίφθη 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 153 καταπίπτει 101 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 155D δέλτα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 110 112 114 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται εγκρίνονται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 καταπίπτει 156 ονομαστικά Πέρας. Απερίφθη. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 149 ονομαστικά. Και πέρας. Απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής ονομαστικά. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ο κύριος Φλέκενστάιν τώρα, εισηγητής. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 2 του κανονισμού παρακαλώ να αναβληθεί η τελική ψηφοφορία. Επί τη βάση εντολής που εγκρίναμε τώρα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως οι δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το αίτημα λοιπόν του εισηγητού ονομαστικά και πέρας. Εγκρίνεται. Αναπέμπεται λοιπόν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να ξεκινήσουν οι δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και περνάμε στην έκθεση Γκουαλτιέρη με την πρώτη ομάδα, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην πρόταση της Επιτροπής, γιατί το δεύτερο μπλοκ καταπίπτει. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Έκθεση για βόρ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Δύο τμήματα. Μονομαστική κλίση το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Παράγραφος 29. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 31. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Παράγραφος. Δύο τμήματα. Ονομαστική και κλίση. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. Ήταν σαφές, αλλά για να είστε ευχαριστημένοι θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Α, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Τι είπα, απορρίπτεται. Ναι, δύο φορές ήρθωσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Προχωράμε στην τροπολογία 6D. Ονομαστική κλίση. Τέλος. Απορρίπτεται. 7D. Με ονομαστική κλίση έρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11, 12, ε, με υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ Α, θέλετε να ελέγξουμε τη 13 Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 13 Τέλος ψηφοφορίας Εγκρίνεται Προχωράμε στην 14 Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 76 ονομαστική ψηφοφορία ε, έρχεται πέρας εγκρίνεται το ψήφισμα με ονομαστική κλίση Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μίλνερ. Μίλναρ. Τροπολογία 4. Αναλλακτικό ψήφισμα. Ε, πρόταση ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά θα το ελέγξω εγώ η ίδια γιατί δεν είμαι βέβαια. Δεύτερο τμήμα λοιπόν, η ονομαστική κλίση, τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παράγραφος 7, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, μονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ αποχές εγκρίνεται. Α, θα το ελέγξουμε. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. τοπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται. Τέλος προφορίας. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 3 σε 3 τμήματα. Συγγνώμη, 10 είναι σε 3 τμήματα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Α, να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Ονομαστική κρίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Άρχεται. Και τώρα τέλος της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές.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 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα της παραγράφου 18. Άρχεται τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Και τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. με πρώτο τμήμα μάλλον, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Πρώτο τμήμα είναι με ονομαστική κλίση. Άρχεται τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 33. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλω να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. Δεν κατάλαβα ακριβώς το αποτέλεσμα. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Υπέρ για του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3. Ε, υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος... Α, να ελέγξουμε για την τροπολογία 3. Μάλιστα, άρχεται. Παρακαλώ να σηκώνετε πιο ψηλά τα χέρια σας. Ε, τέλος ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Εγκρίνεται, συνάδελφοι. Και περνάμε στην παράγραφο 36, με ονομαστική κλίση, άρχεται. Και τώρα Τέλος, εγκρίνεται. Εκτιμώντας 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 1. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική σκέψη α, ονομαστική κλίση, άρχεται, τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική β, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σ, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας οι δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική F, ονομαστική κλίση, άρχεται, τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική H, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική L, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά τέλος πληροφορίας εγκρίνεται λοιπόν ε, ε λογική π πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αιτιολογική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική τα υπέρ, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική W με ονομαστική κλίση άρχεται τέλος και εγκρίνεται. Αιτιολογική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική Z πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. And the vote is now closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνάδελφε, περνάμε στην έκθεση Honeyball. Ξεκινάμε με την τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα κάνουμε όμως έλεγχο. Ανοίγει η ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέραγραφο 1 από το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Τον κάνετε. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Μάλλον άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. γίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Πέρασμα, μάλλον. Παράγραφος 2 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρασμα. Εγκρίνεται. παράγραφο 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Με ονομαστική ψηφοφορία μάλλον. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. δεκατρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δεκαπέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την πρώτη τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Δεν είναι σαφές. Δεν την άνταση Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 26 τα πιπτή. 29 σε 4 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές αγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές αγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές αγκρίνεται. Παράγραφος 32 πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, 31. Άρχεται ψηφοφορία για τα 31. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφος 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία έρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία μάλλον. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα μάλλον υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 37 ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρα. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν κρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Είναι μαστική ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 40, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 42, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 43. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ονομαστική μάλλον ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 50. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 ονομαστική πληροφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Όλες οι ηλεκτρονικές. Πρώτο βήμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία περάσω. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρασε. Δεν κρίνεται. Ρίσα τα λτζή. Επιλογή και το Υπέρ. Κατά. Αποχέ. το Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν κρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν κρίνεται. Επιλογική σκέψη ήταν H. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Recital P. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ετεολογική σκέψη Α. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Ετεολογική σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Ετεολογική σκέψη W υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τέλο ψήφισμα συνολικά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλιστα. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Μια διακοπή πριν περάσουμε στις εξηγήσεις ψήφου. Καλή όρεξη. Συνάδελφοι, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε τις εξηγήσεις ψήφου, οπότε παρακαλώ όσοι δεν συμμετάσχετε να βγείτε από την αίθουσα.